συνεδρίαση στις Παρασκευή 24ης Απριλίου έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά. Δεν υπάρχουν. Θεωρείται λοιπόν ότι κυρώνονται, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Ο συνάδελφος Μπλόκλαντ ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Μπλόκλαντ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε είναι ένα, μια επέτειος ετήσια, μια γιορτή στην Ολλανδία η μέρα της Βασίλισσας με την οικογένεια του βασιλικού οίκου της Οράγγης. Εξακολουθούμε να ε, βρισκόμαστε υποκαθεστώς δέους για όσα συνέβησαν και για τα συλληπιτήρια ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την επιστολή που απεστάλλει στη Βασίλισσά μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε Μπλόκλαντ, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, για την απόφαση της 30 Απριλίου 2009 το 10 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση σε 393 κάθετος 07 Ιταλική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην υπόθεση σε 9 κάθετος 08 Μπενιαμίνο Ντονίτσι κάθετος Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε την εξής νομολογία. Αναφέρω, η απόφαση 2007 κάθετος 212 REG ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2007 για τον έλεγχο της εντολής ε, του Μπενιαμίνο Ντονίτσι θεωρείται άκυρη. Τέρμα παραθέματος. Τέλος